Λοιπόν, τα πρακτικά αυτά της συνεδρίασης. Δύο ομάδες, και και έχουν υποβάλει προτάσεις για την ένταξη στις αντιπροσωπείες. Ευρωμέτα Σιάν, ο κύριος Στάκουλα, αντί της κυρίας Στάινεν. Ο κύριος Μιλάνα, αντί της κυρίας Μπαλσάνη. σχέσει με τι χώρε της Νότια Ασίας. Βαρτσάνη αντί Μιλάνα. Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Κόβαλ αντί του κυρίου Σιμάνσκι. Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμηνίας Σιμάνσκι αντί του κυρίου Κόβαλ. Διαφωνεί κανένας με τις αλλαγές αυτές. Δεν βλέπω. Εγκρίνω λοιπόν οι ορισμοί αυτοί. Σύμφωνα με την διάταξη, περνάμε τώρα στην κοινή συζήτηση για τη δήλωση τη Κομισιόν και του Συμβουλίου για τη Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση Τατζικιστάν και τη